Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ όλους τους εδώ παρόντες. για τι προσπάθειε που για να έρθουν εδώ. Ξέρετε ότι είχαμε πολλέ δυσκολίε να φτάσουμε μέχρι το Στρασβούργο. Πολλοί συναδελφοί δεν τα κατάφεραν μάλιστα. Μόλι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση τη διάσκεψη των Προέδρων, των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένε προτάσει να υποβάλουν στο σώμα. προτάσει τι οποίε υποστηρίζουν ομόφωνα οι Πρόεδροι των Πολιτικών Ομάδων και σα τι ε, ε, αναφέρω. Συνοπτικά θα σας πω ότι προτείνουμε να μην γίνει η συνεδρίαση της Ολομέλειας την Πέμπτη. Δεν θα υπάρξει δηλαδή μέλη συνέντευξη για την Πέμπτη. Ταυτόχρονα όμως μπορείτε την Πέμπτη το πρωί να υπογράψει στον κατάλογο των, των παρόντων και ο κάθε βουλευτής μεμονωμένα μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του ενδεχομένως. Αλλά πάντως σύνοδος Ολομέλειας δεν θα γίνει. Η δουλειά πρέπει να συνεχίσει, είναι καθήκον μας. Όποιο λοιπόν υπογράψει τον κατάλογο παρουσιών την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα θεωρηθεί ότι όντω ήταν εδώ παρόν και εργάστηκε όπω πάντοτε, δεν υπάρχει δηλαδή διαφορά. Αυτή την εβδομάδα επίση θα πρέπει να σα πω ότι δεν πρόκειται να γίνουν ψηφοφορίε ούτε κατά την Ολομέλεια ούτε κατά τι συνεδριάσει των Επιτροπών, εφόσον έχουν προβλεφθεί συνεδριάσει Επιτροπών, οι οποίε δεν μπορούν να λάβουν χώρα, αλλά και μάλιστα ακόμη και την Πέμπτη, εάν μια Επιτροπή στήσει να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, δεν υπάρχει αντίρρηση, χωρί όμω ψηφοφορίε. Και αυτό είναι η απόφαση που λάβαμε, διότι διαπιστώσαμε ότι πολλοί συναδέλφοι για λόγου πρακτικού δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατή δηλαδή η μετάβασή του στο Στρασβούργο και δεν μπορούμε να του αποστερήσουμε το δικαίωμα τη συμμετοχή σε αυτή την σύνοδο. Δεν τίθεται ζήτημα δηλαδή βεβαίω απαρτία, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει απαρτία. Απλώ σεβόμενοι το γεγονό ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν να φτάσουν μέχρι το Στρασβούργο, δεν θα πραγματοποιήσουμε ψηφοφορίε. Η αναβολή των ψηφοφοριών όμω δεν θα έχει ε, επιπτώσει ω προ τι ε, υποχρεώσει μα τι ε, νομοθετικέ εναντί του Συμβουλίου. Αναβάλλονται κατά δύο εβδομάδε οι ψηφοφορίε και θα λάβουν χώρα κατά την Ολομέλεια που έχει προβλεφθεί για τι Βρυξέλλες σε δύο εβδομάδες. Και η διαδικασία συνεργασία με το Συμβούλιο και η διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης θα τηρηθούν όπως πρέπει. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ε, πληροφορία που θέλω να σας ανακοινώσω και επίσης θα θέλω να σας ενημερώσω ότι για λόγους πολύ σημαντικούς γίνεται η σημερινή συνεδρίαση γιατί προβλέπεται για αύριο ένα σημείο έκτακτο που δεν είχε ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη μέχρι τώρα. Ένα σημείο που έχει να κάνει με, την, με τα προβλήματα στην ενέργεια κυκλοφορία στην Ευρώπη και τα προβλήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Βλέπετε λοιπόν μια συνεδρία σε αύριο δύο ωρών, παρουσία και του Πρόεδρου Μπαρόσο. Θα συζητήσουμε δηλαδή την κατάσταση στην Ευρώπη, τα προβλήματα στις μεταφορές, μετακινήσεις, που έχουν όπως ξέρετε ε, περιοριστεί ιδιαίτερα που ενδέχεται και να προκαλέσουν ε, σημαντικά προβλήματα απασχόλησης στις ε, μεγάλες, στα μεγάλα αεροδρόμια και τις μεγάλες αεροπορικές επιχειρήσεις εκ των οποίων ορισμένες κινδυνεύουν και με πτώχευση ακόμη λόγω αυτών των μεγάλων προβλημάτων στις ενέργειες μεταφορές. Έχει τεράστια σημασία αυτή η συνεδρίαση αύριο λοιπόν. Και ενώ δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική ημερήσια μας διάταξη, σημειώσαμε, συμπεριλάβαμε και το θέμα αυτό, διότι αναγνωρίζουμε τη μεγάλη, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενανερείς μεταφορές στην Ευρώπη και πρέπει αναγνωρίζουμε να τα συστήσουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Κάποια άλλα θέματα ενδεχομένως να συζητηθούν και για την Πέμπτη αύριο 9 το πρωί. Σε, σε μερικά λεπτά θα σα εξηγήσω τα πάντα. Μέρα, μέρα τη μέρα θα σα εξηγήσω την ημερήσια διάταξη. Μόνο κάποιε γενικέ πληροφορίε θα σα δώσω. Και προχωρώ. Για να σας ε, καταστήσω γνωστό ότι στις 7 Απριλίου έλαβα επιστολή του κυρίου Φάρετζ, συμπροέδρου της Ομάδας Ευρώπη και Δημοκρατίας καλείται το σημείο 6 του κανονισμού, το άρθρο 6 μάλλον, και ε, διαμαρτύρεται ε, για τον τρόπο ε, με τον οποίο χειριζόμαστε στην Ευρώπη